και οι αρμόδιες Ιταλιακές αρχές ε, του κ. Μαζελίνη θα, ε, θα είναι υπό την ηγεσία του κ. Ζαλίνη μετά τον κ. Λούπι. Ο κ. Ζαν Ποντάν μετά την ε, πρώτη συνεδρίαση της, του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης ό,τι αφορά, ενημερώθηκε το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την εκλογή του κυρίου Φιλίπ Λουαζό. Και σύμφωνα με το 7.1 της πράξης για τις άμεσες εκλογές ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με το 1 και 4 του κανονισμού, το Κοινοβούλιο αποδέχεται την εκλογή του κυρίου Ζαλίνη και του κυρίου Λουαζό από 1η Ιουλίου 2014. Καλώς ορίζω λοιπόν τους καινούριου συναδέλφους και να σας επενθυμίσω ότι σύμφωνα με το 3-2 του κανονισμού έχουν πλήρη δικαιώματα και μπορούν να συμμετάσχουν, να συμμετέχουν ε, στη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου και δεσμεύονται γραπτά ότι δεν υπάρχει αντιφατική θέση την οποία ανακατέχουν σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή ως βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προτάσεις στη διάσκεψη των Προέδρων για τον διορισμό στις Επιτροπές ε, υποβλήθηκαν χθες και δεν υπήρξαν τροπολογίες που να κατατέθηκαν. Άρα, σύμφωνα με το 1919-3 του κανονισμού, θεωρούνται ότι εγκρίνονται αυτές οι προτάσεις. Τα πρακτικά αυτές τις συνεδρίασεις θα ζητηθούν κατά την επόμενη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου προς έγκριση. Από την δικιά σας πλευρά υπάρχει κάποια παρατήρηση για κάποια από αυτά τα θέματα. Όχι. Τότε λοιπόν διακόπτεται η συνεδρίαση πέρα τη συνεδρίαση.